Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, είμαστε υποχρεωμένοι στην επανάληψη έναρξη μιας συνόδου να αναθυμηθούμε και να μνημονεύσουμε αθώα θύματα. Θύματα της παράλογης μανίας της τρομοκρατίας. Μια πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λονδίνο, πλήγει με πολλά θύματα από διάφορες εθνικότητες. Όμως ε, η φωνική τρομοκρατία χτύπησε και εκτός σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίθεση στη Βουλή της Τεχεράνης που δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε είναι και αυτή μια φρικτή επίθεση. Γνωρίζουμε ότι η δύναμη της ελευθερίας και της δημοκρατίας δεν θα λυγίσουν μπροστά στο φόβο της βίας, της τρομοκρατίας. Δεν θα αλλάξουμε το δικό μας τρόπο ζωής. Θα προχωρήσουμε ως Ευρωπαίοι και θα δώσουμε μια αποφασιστική συμβολή στην προσπάθεια να ιτηθεί η τρομοκρατία. Πέραν αυτού όμως, θα σας καλέσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Λονδίνου και της Τεχεράνης. Συνάδελφοι, πρώτο και ρίξω την έναρξη της Συνόδου να εκφράσω και την ανησυχία μας για την τύχη του δικηγόρου Τάνερ Κίνιτ, του διευθυντή τη ε, Διεθνού Αμνηστία στην Τουρκία, ο οποίο συνελήφθη από τι τουρκικέ αρχέ την περασμένη Τετάρτη μαζί με άλλου 22 δικηγόρου. Ζητούμε από τις αρχές της Τουρκίας την άμεση απελευθέρωση του Τάμερ Κίριτς και όλων των υπολείπων που συνελήφθησαν και να ε, ανακληθούν όλες οι κατηγορίες εναντίον τους, προτού βρεθούν σαφή υποδεκτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ε, την ανάμεξή τους στην αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016. Επίσης, θέλω να θυμίσω ότι η Ευρώπη είναι μια κοινότητα αξιών και ελευθεριών και ότι πάντοτε θα είμαστε στο πλευρό όλων όσοι μάχονται για να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη έχει αναλάβει να υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό θέλω να εκφράσω ξανά την ανησυχία μας σε σχέση με τη σύλληψη σήμερα το απόγευμα του αρχηγού της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέη Ναβάλνη και άλλων υποστηρικτών του που βρίσκονταν μαζί του. Να μην ξεχνάμε ότι όπως και σε άλλες περιπτώσεις τα θύματα βίας και διακριτικής μεταχείρισης πρέπει να μνημονεύονται. Ε, θα πρέπει λοιπόν να θυμίζουμε την κοινότητα αξιών που συμμεριζόμαστε και προσπιζόμαστε και των οποίων είμαστε άοκνοι υπερασπιστές. Θέλω να τονίσω και ότι ο κύριος Γιαζίν Αλτολούλ, ο οποίος συνελήφθη στο, σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, η κυρία μάλλον, ε, απελευθερώθη χωρίς καμία κατηγορία εναντίον της. Κυρίσω την επανάληψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί στην, ε, την Πέμπτη 18 Μαΐου. Τα πρακτικά από τις προηγούμενες συνόδους είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Τα πρακτικά θεωρούνται